που ζητούμε. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις πρωτοβουλίες στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, τόσο ώστε να σημειωθεί πραγματική πρόοδος. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Σλίτερ. Ε, και τώρα ακολουθεί ε, ο κύριος Σεγγεντή.